Do you know which seat we are? Uh, I think it's Because it so. Right, good, good morning. Um, I think they'd uh, not... Καλημέρα. Είχαμε ένα προβληματάκι με τις θέσεις και τα μικρόφωνα, αλλά διορθώθηκε λοιπόν. Θα εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη. Φαντάζομαι ότι δεν έχει κανείς αντίρρηση. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Πρώτο δε θέμα είναι το δικό μου. Θα πάρω λοιπόν μόνη μου το λόγο για να σας εξηγήσω τι λέει η έκθεσή μου. Σας υπενθυμίζω ότι οι συντονιστές μου ζήτησαν να το κάνω γιατί είχα κάνει πολλές εκθέσεις αναχώρα χώρα και άρα μου έδωσαν και την εντολή να είμαι όσο το δυνατόν αυστηρότερη και σκληρότερη. Ελπίζω λοιπόν συνενετικά να με βοηθήσετε και για τις τροπολογίες όταν θα έρθει η ώρα τους, αν έχετε κι εσείς καμιά ιδέα. Η Κομισιόν έκανε την πρότασή της σε περίεργη εποχή, διότι μόλις δημοσιεύτηκε εγκρίθηκε η Οδηγία Λογιστικών 2013 που αντικαθιστούσε τις προηγούμενες και βασιζόταν σε αυτές, τροποποιώντας τις. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να πούμε ότι τροποποιούμε κάτι που δεν υπάρχει πια και άρα οι όλες οι τεχνικές αλλαγές για τις τροποποιήσεις του ανύπαρκτου πλέον αυτού πράγματος είναι η Λογιστική Οδηγία 2013. Μπορεί λοιπόν να ανοίγουμε μια υπόθεση που έχει οριστικά κλείσει. Είπαμε να μην το κάνουμε για να μην διαταραχθεί η ισορροπία. Είπε λοιπόν η Κομισιόν να δίνονται περισσότερες πληροφορίες από τις εταιρείες στο κοινό όπως περιβαλλοντολογικά και εργασιακά θέματα, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και καταπολέμηση της διαφουθοράς. Και αν δεν το πράξουν τότε θα πρέπει να εξηγούν και γιατί. Τρία κύρια θέματα έχει η έκθεσή μου οι εκθέσεις χώρα με τη χώρα, ο σχεδιασμός των φορολογικών μέτρων και το θέμα αυτό της πληροφόρησης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Καταρχήν λοιπόν χώρα με χώρα. Από την, λογιστική, από την συμπλήρωση της λογιστικής συμφωνήθηκε από τα συμπαράσματα του Συμβουλίου των Μάιων να, επεκταθεί, να επεκταθούν οι εκθέσεις αναχώρα. Δεν είμαι βέβαιη ότι γνώριζαν ακριβώς τι εννοούσαν, αλλά αυτό είπανε. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε τέτοιου είδους αναφορές. Πολλές φορές μας λένε ότι οι αναφορές χώρα με τη χώρα μπορεί να είναι κάτι το αρνητικό και γι' αυτό έβαλα τη ρήτρα ότι αν είναι αρνητικό να μπορεί να αλλάξει και αντί να δημοσιεύεται ευρέως να πηγαίνει μόνο στις φορολογικές αρχές. Θα ζητήσω από τη γραμματεία να το ψάξει για το νομικό υπόβαθρο. Είναι ο φόρος η βάση ίσως να πρέπει να τα υποβάλουμε όλα αυτά και αλλού, όχι μόνο στις φορολογικές αρχές. Λέω λοιπόν, θα φροντίσω όλα να συμφωνούν με το άρθρο 114. Ακούω ακόμη ιδέες ως προς το σωστότερο τρόπο για να τα κάνουμε όλα αυτά. Αν έχετε ιδέες να τις ακούσω. Εγώ τροποποίησα το κεφάλαιο 10 της Λογιστικής Οδηγίας 2013 που ορίζει για πρώτη φορά τι είναι η αναφορά χώρα με χώρα, χώρα τη χώρα και το έβαλα εκεί γιατί ήθελα να υπάρχει και δημοσιονομικός έλεγχος και έλεγχος αυτής της πληροφόρησης γιατί μερικοί είπαν αν τα βάλουμε στην ετήσια έκθεση τότε είναι υπερφορτωμένοι αλλά εγώ νομίζω ότι αν έχετε άλλες ιδέες να τις ακούσω. Πρέπει όμως νομίζω να υπάρχει κάποια διαβεβαίωση ότι όλα αυτά θα συμφωνούν με τις δημοσιονομικές δηλώσεις. Το δεύτερο, η ευθύνη. Αυτό δεν είναι οριζόντιο θέμα, αφορά χρηματοπιστωτικά ιδουρήματα. Και εδώ λέω ότι λόγω της κυριαρχίας του δημοσιονομικού συστήματος στο σύνολο της οικονομίας μοιάζουν όλα αυτά λίγο με τις διατάξεις για τις δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεων. Γι' αυτό αυτή την έννοια την έβαλα και αυτή στην έκθεσή μου ελπίζοντας να εφαρμοστεί με τη ρήτρα αυτή τη ειδική ευθύνη, δηλαδή πληροφόρηση για την εκπαίδευση του προσωπικού και της διαμεσολαβήσεις με στόχο να βελτιωθούν οι σχέσεις, οι εργασιακές σχέσεις της εταιρείας. Επίσης, έβαλα πρόσθετες, ε, πρόσθετη πληροφόρηση για να υπάρξει κάποια αναλογικότητα με τις μεθόδους επιθετικών μειώσεων φορολογίας ανάλογα με τις συμβουλές που παίρνουν οι εταιρείε από εξωτερικούς συμβούλους. Και αυτά συμφωνούν και με τη δουλειά του ΟΣΑ, του ΣΥΤΑ 20 και της Κομισιόν που στοχεύει στην μείωση των φορολογικών παραδείσων. Θεώρησα ωφέλιμο για τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν γενικά κανόνες anti-avoidance που εφαρμόζονται ήδη σε πολλές χώρες εκτός Ένωσης είπα Νότια Αφρική, Καναδά, Αυστραλία και Χονγκ Μόγκ και αρχίζει να εφαρμόζεται και στο ΙΤΑΒ. Άλλες αλλαγές το εύρος στο πεδίο εφαρμογής εδώ κοίταξα τι απαιτεί η οδηγία και ποιες ε, εταιρείε καλύπτει. Οποιαδήποτε λέει η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση με 500 ή παραπάνω υπαλλήλους με ισολογισμό πάνω από 20 εκατομμύρια ή τζίρο 40. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται αυτά τα διπλά κριτήρια, διπλά όρια, γιατί οποιαδήποτε ευρωπαϊκή εταιρεία που έχει τέτοιο ισολογισμό και τζίρο είναι ούτως ή άλλως υποχρεωμένη να δίνει αυτές τις πληροφορίες ανεξαρτήτως από το πόσους απασχολεί. Γιατί τέτοιου είδους ισολογισμοί έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομία των χωρών όπου εργάζονται, όπου λειτουργούν. Η προσέγγιση της Κομισιόν είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι οι εταιρείε πρέπει να αποδεικνύουν πώς κατέληξαν στις, στα προγράμματα που εφαρμόζουν σε περίπτωση καταστροφών όπως στην Μπαγκλαντές όπου φαίνεται ότι μπορεί οι ζημίες να είχαν μειωθεί αν είχε υπάρξει ιδέουσα επιμέλεια. Due diligence το λένε οι δήμονες. Για τα υπάρχοντα πλαίσια η πρόταση της Κομισιόν αναφέρεται σε εθνικά προγράμματα και σε αυτά που εφαρμόζουν οι μεγάλες ενωσιακές επιχειρήσεις. δεν υπαγορεύει τα πάντα, όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να το κάνουν, αλλά κάτι τέτοιο πρέπει να εφαρμόζουν για να αναγνωρίζονται οι κατευθυντήρες κύριες ιδέες αυτών των πληροφορήσεων και από τους ενδιαφερομένους. Με συγχωρείτε γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές μου τροπολογίες Ίσως να μπορέσουμε να τις βάλουμε όλες μαζί σε, έναν κολοσιαίο, για μια κολοσιαία συμβιβαστική. Και βέβαια αν η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν τα κάναμε σωστά να μας το πει και να τα προσαρμόσουμε. Αλλά έκανα διαβουλεύσεις και νομίζω σωστά τα είπα. Αυτά είναι βασικά, αυτό είναι βασικά το περιεχόμενο της εκθεσής μου και θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης και πρώτο πρώτο το Ζαν Πολ. Λοιπόν, βρήκα και ένα μικρόφωνο που δουλεύει, επομένως μπορώ να πάρω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να ακρηγορήσω γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας και ε, ξέρω ότι είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να πάρουν το λόγο για αυτό το συγκλονιστικό θέμα. Θα πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την έκθεσή σας, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη αντίρρηση. Με προβληματίζει λίγο το θέμα της συνοχής, δηλαδή η συνεκτικότητα μάλλον με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα για τις εταιρείε. Νομίζω ότι καλό είναι που θέλουμε να ρυθμίσουμε περισσότερο, καλό είναι να τακτοποιήσουμε τα πράγματα, να βάλουμε τάξη, αλλά όχι ε, αυτό να αποβεί σε ζημία της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν οι απαιτήσει ε, να είναι χρήσιμες και ωφέλιμες. Δεύτερον, ε, καλό είναι να έχουμε απαιτήσει. Όμως, εάν δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πραγματικότητα των δραστηριοτήτων, τότε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Διαπιστώνουμε ότι δίνουμε μεγάλες αρμοδιότητες πλέον σε διάφορους οργανισμούς ή υπηρεσίες, π.χ. χρηματοοικονομική εποπτεία κτλ. Χωρίς όμως να τους δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία ε, χρηματοπιστωτικά και άλλα για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Επομένως, δεν θα ήταν καλό να βαρύνουμε τις ε, επιχειρήσεις ε, με επιπλέον διοικητικό άχθος. Θα πρέπει να στοχεύουμε μόνο στα ουσιώδη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι καλά ζυγισμένες αυτού του είδους οι νομοθεσίες. Και να πω ότι αν υπάρχει απάτη εντάξει, αλλά εάν υπάρχει ε, φόρο διαφυγή, ε, ε, εκεί ευθύνονται τα κράτη. Είναι λογικό ο φορολογούμενος να προσπαθεί να πληρώσει όσο γίνεται λιγότερο στην εφορία, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι χώρες, τα κράτη μάλλον είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να προσέχουν, να μην δίνουν πολλές οδούς διαφυγής σε αυτούς που δεν θέλουν να πληρώνουν ε, το, τους φόρους τους. Επομένως, οι φορολογικές αρχές ε, είναι αυτές των κρατών μελών, ε, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα, τα οποία να εφαρμόζονται εύκολα, αλλά και ο έλεγχος τους να είναι εύκολος και ευχερής. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Δεν ξέρω μήπως μπορούν να βοηθήσουν λίγο οι τεχνικοί, αλλά έχουμε πρόβλημα μεγάλο με τα μικρόφωνα. Δεν δουλεύει κανένα. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Ναι, πρέπει κάτι να γίνει, γιατί διαφορετικά θα παίζουμε όντως μουσικές καρέκλες εδώ, θα ψάχνουμε... Λοιπόν, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να στηρίξω την έκθεση της ε, Προέδρου γιατί είναι πάρα πολύ σωστή και μπορώ να συμφωνήσω με πάρα πολλά από τα σημεία τα οποία αναφέρει και επί της αρχής και επί της ε, ουσίας. Ε, όσον αφορά ε, το θέμα αυτό και η αναφορά χώρα-αναχώρα είναι πολύ σημαντική. Πάντως προτείνουμε το άρθρο 42 να παραμείνει ε, απαράλλακτο. και η πρόταση που κάνετε για το άρθρο αυτό να συμπεριληφθεί σε μία άλλη, σε μία άλλη τροπολογία. Να συνεχίσει η ομιλήτρια παρακαλώ. Λοιπόν, συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αλυσίδα ε, τροφοδοσίας, όμως Ξέρουμε όλοι τι, συνέβη στον Μπαγκλαντές, ε, ξέρουμε τέτοια προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια και συμμόρφωση προς τους κανόνες. Δηλαδή ή θα πρέπει να συμμορφούνται ε, οι ενδιαφερόμενοι ή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν την ε, θέση τους ή την κατάσταση. Αυτό σημαίνει διαφάνεια. Ε, έχει υπογραμμιστεί το θέμα στην έκθεση, το θέμα της επιθετικής φορολογικής πολιτικής. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ενδεχομένως, εάν πιέσουμε πάρα πολύ, μπορεί να δημιουργήσουμε προβλήματα σε επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν καλά, νόμιμα ε, και επομένως ε, ε, κάνουν νόμιμα κέρδη, παράγουν νόμιμα κέρδη. Να μην βαρύνουμε αυτές τις εταιρείες. Επομένως, ναι, ένας σωστός, μετρημένος, ζυγισμένος βαθμός επιθετικότητας για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα σε επιχειρήσεις. Όσον αφορά την τροπολογία 28, να πω το εξής. Προσπαθεί η έκθεση να εξηγήσει τι γίνεται με τις μικρές επιχειρήσεις ε, και γίνεται μια ε, προσπάθεια ε, να απαλληφθεί ο αριθμός των εργαζομένων και για τον τζίρο, για τον κύκλο εργασιών θα δούμε αν θα μείνει στα 20 ή στα 40 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι είναι σημαντικός ο αριθμός των εργαζομένων της μικρομεσαίας επιχείρησης. Όμως με τον αριθμό των εργαζομένων ε, κανονίζουμε το εάν είναι μικρομεσαία η επιχείρηση. Επίσης πρέπει να δούμε αν δουλεύει σε εθνικό ή ε, διεθνές πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να επιλεγεί πάντως ένα πλαίσιο. Αυτά είχα να σας πω να πω για μία ακόμα φορά ότι είναι εξαίρετη η έκθεση και βεβαίως ε, μπορούμε να την στηρίξουμε με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα γίνουν σεβαστές και οι δικές μας τροπολογίες. Ε, από τους Πρασίνους, ο κύριος Λάμπερτς. δουλεύει το δικό μου μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Ε, το βρίσκω λίγο περίεργο να πω την αλήθεια, γιατί έχουμε μια φιλελεύθερη συγγύτρια που λέει ναι αυτό πρέπει να το κάνουμε και οι εταιρείε ε, μπορούν να τα κάνουν αυτά χωρίς προβλήματα και ο Ζαν Πολ και κάποιοι σοσιαλιστές λένε όχι ναι να είμαστε λίγο συνετοί τι συμβαίνει εδώ κάθε φορά που κάνει η Σάρον μια έκθεση αισθάνομαι ε, και πιο φιλελεύθερος περίεργα πράγματα τέσσερα είναι εξαιρετική η έκθεση Ζαν Πολ Λοιπόν, όταν λες, ε, Ζωάν Πολ, ότι πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να μην ε, ε, επιβάλλουμε ιδιαίτερες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, συμφωνώ. Αλλά και εγώ έχω δουλέψει σε, μεγάλες, σε μια μεγάλη επιχείρηση όπως και εσύ. Αλλά ξέρετε ότι δεν χρειάζεται τώρα να τις φτιάξουν για μας αυτές, αυτούς τους λογαριασμούς και αυτά τα στοιχεία οι μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουν τα στοιχεία αυτά ήδη. Επομένως, πρέπει να δούμε εάν πραγματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν έχουν αυτή την ικανότητα. Αυτό που είπε η Σάρων είναι λογικό. Δηλαδή κυρίως τα νούμερα του τζίρου και του ισολογισμού έχουν σημασία. Μπορεί να βγάλει κανείς πολλά λεφτά με λίγους υπαλλήλου τώρα πια. Οπότε, για το οικονομικό κομμάτι των μη οικονομικών αναφορών μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση τριπλή, δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιρούνται, οι μεγάλες ε, υπάγονται και στο ενδιάμεσο θα υπάρχει συμμόρφωση ή εξήγηση. Να έχουμε δηλαδή μια, φάση, μια προσέγγιση τριών ε, επιπέδων για να μην ανησυχούν και οι άλλοι συναδελφοί ότι υπερφορτώνουμε τις χώρες. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τις μεγάλες εταιρείες ανά χώρα και μετά θα δούμε πώς θα το επεκτείνουμε σε περισσότερες εταιρείες. Αλλά ας προσπαθήσουμε πρώτα να πιάσουμε τα μεγάλα ψαριά. Όσον αφορά τώρα την, ε, τα θέματα ανταγωνισμού και ε, φοροαποφυγής, ε, ναι, βεβαίως συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν, να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι μας ενδιαφέρει το κέρδος, όχι, μας ενδιαφέρει μόνο η μη συμμόρφωση με τους φορολογικούς νόμους. αλλά πώς να σας το πω, τα κράτη δεν θέλουν πάρα πολύ αυτήν την την διαφάνεια που θέλουμε εμείς στο Κοινοβούλιο να πιέσουμε πολύ όσον αφορά ε, την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Εμείς ε, πρέπει να πιέσουμε ε, και τις χώρες και αυτό άλλωστε κάνει το reporting αναχώρα. Επομένως, εάν έχουμε τα στοιχεία και αν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, τότε κατά κάποιο τρόπο θα πιεστούν και οι ίδιες οι χώρες έτσι ώστε ε, να ε, επιτύχουν ένα βαθμό ε, συγκρισιμότητας. Νομίζω ότι τώρα στις 28 χώρες, εάν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία διαθέσιμα, τότε θα είναι εύκολο για τις επιχειρήσεις. Θέλω επίσης να τονίσω κάποια άλλα θέματα για την αλυσίδα της ε, αξίας. Ε, το έχει εξηγήσει αυτό Σάρον σε ένα εκτιμώντας. Αναρωτιέμαι πώς πρέπει να μπει σε άρθρο και να πούμε πώς υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις τουλάχιστον για μεγάλες εταιρείε όσον αφορά τουλάχιστον ε, το να αναφέρουν την αλυσίδα δημιουργίας αξίας και νομίζω πως πράγματι θα δημιουργηθεί έτσι περισσότερη πειθαρχία για την αναφορά του κινδύνου τώρα. Θεωρούμε πως πρέπει να φροντίσουμε να καλύπτουμε κάθε είδος κινδύνου και μετά την κρίση του 2008 ασχολούμαστε με τον οικονομικό κινδύνο, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη κινδύνου. Διαχείριση κινδύνου, αξιολόγηση κινδύνου βεβαίως δεν είναι κάτι το ακριβές, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό οι χώρες να αξιολογήσουν ε, τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Φανταστείτε, ξέρω εγώ, μέρος της αλυσίδας παραγωγής να είναι στην Τινησία ή στην Αίγυπτο. Ειδικά στε... αν φτιάχνει κάποιος ρούχα. Ε, και να ξεσπάσει η Αραβική Άνοιξη. Πρέπει λοιπόν να το δουν και από πλευράς ε, γεωγραφίας και γεωπολιτικής. Το μέτωπο αυτό κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Πρέπει να καλύψουμε λοιπόν και αυτές τις πτυχές. Τι άλλο. Αυτά νομίζω. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη βασική εκθέση. Θέλουμε να τη βελτιώσουμε λίγο, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν υπάρχουν και πολλά να βελτιώσουμε. Σας ευχαριστούμε Φιλίπ. Δεν είναι εδώ ο Άσλι. Α, εδώ είναι, συγγνώμη. Ναι. Έχεις το λόγο. Σε ευχαριστώ Σάρα. Η πρόταση αυτή δεν διαφωνεί με ό,τι ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και γι' αυτό δεν έχω κι εγώ σημαντικές αντιρρήσεις. Άκουσα αυτά που είπε ο Ζαν Πολ για τα βάρη που θα χρειαστεί να φέρουν περαιτέρω οι επιχειρήσεις. Και δεν πρέπει να τις επιβαρύνουμε πολύ. Εκτιμώ τις προσπάθειές σας να χτενίσετε το κείμενο και να ευθυγραμμίσετε την υποχρέωση αυτή πληροφόρησης και με άλλη νομοθεσία. Και συμφωνώ επίσης να είναι κύριο κριτήριο ο τζίρος και όχι ο αριθμός των ε, υπαλλήλων θα ήθελα να μειωθεί το εύρος και να καλύπτει μόνο τις εταιρείε των οποίων οι μέτοχοι θα ωφεληθούν από αυτές τις πληροφορίες. Επίσης οι αναφορές χώρα με χώρα με βρίσκουν σύμφωνο και δεν θα ήθελα να προωθήσουμε πρωτοβουλίες που μπορεί τελικά να βλάψουν τις επιχειρήσεις. Okay, thank you very much. Is there anybody else wanting to come in? Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Δεν βλέπω κάποιον. Όλοι καφέ θέλουν. Κανείς δεν θέλει να μιλήσει. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Αναμένω τις ε, τροπολογίες. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να συμπεριλάβω αυτές ε, που θεωρώ πως ταιριάζουν με τη γενική ιδέα ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε περισσότερη διαφάνεια για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Είναι θέμα που ανησυχεί ιδιαίτερα την κοινή γνώμη τη στιγμή που πάρα πολλά κράτη-μέλη θέλουν να αυξήσουν τα φορολογικά τους έσοδα οι μεγάλες εταιρείες φαίνεται πως μπορούν να πηγαίνουν τα χρήματά τους όπου θέλουν και να μην πληρώνουν. Να μην πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί. Και αυτό έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Το έχουμε συζητήσει στο πλαίσιο διαφόρων πραγμάτων. Οικονομική διακυβέρνηση, φόρος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αν είναι να ανακάμψουν τα οικονομικά των κρατών μελών, οι εταιρείε πρέπει και αυτές να υπομιστούν αυτό που τους αναλογεί και βεβαίω οι εκθέσεις αναχώρα, κάτι το οποίο βεβαίω βοηθούσε ανατσόμενες ε, χώρες, ε, φαίνεται πως ε, έχει φτάσει η ώρα να χρησιμοποιηθεί και στον ανεπτυγμένο κόσμο για να μπορέσουμε και εμείς να φορολογήσουμε. Αναμένω λοιπόν τις τροπολογίες. Ε, να δούμε πού θα πάνε τα διάφορα διάφορες διατάξεις στα διάφορα άρθρα. Η Κομισιόν θέλει να μας δώσει και κάποιες, αν θέλει να μας δώσει κάποιες συμβουλές, ευχαριστώ. Και από την ε, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας ε, και Αγοράς, δεδομένου του ότι είναι μια πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς. Ο χρόνος πιέζει, δεν έχω δώσει το χρόνο τον λόγο στην Θέλετε να μιλήσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, το θεωρώ απαραίτητο. Οπότε θα καθίσω εδώ πέρα για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε τις συμβουλές σας, όπως σας είπα μήπως έχουμε ξεπεράσει κάπου την ε, νομική βάση του άρθρου 114. Ε, Οι προθεσμοί για τροπολογίες είναι πολύ πιεστικοί για να τελειώσει εγκαίρως η γνωμοδότηση. Είναι λοιπόν στις 6 Νοεμβρίου η προθεσμία. Μέχρι τα μεσάνυχτα. 21 Νοεμβρίου θα εξεταστούν τροπολογίες και θα ψηφίσουμε. Οπότε ελπίζουμε να έχουμε κάποιες ε, συμβιβαστικές προτάσεις μέχρι τότε. Στην Ολομέλεια δεν έχουμε πάει ακόμα, γιατί η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι η κύρια Επιτροπή. Παρά το ότι βεβαίως σε κάποιους τομείς έχουμε κοινή αρμοδιότητα με άλλες. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Εγώ πρέπει να φύγω. Θα δώσω την προεδρία στον Πάμπλο. Αν βρει ένα μικρόφωνο βεβαίως που δουλεύει. Καλημέρα σε όλους σας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Θα μιλήσω αγγλικά, αν μου το επιτρέπει ο κύριος Γκοζές. Ανακοινώσεις ε, του Προέδρου όσον αφορά τους ε, τριμερείς ε, διαλόγους στήριξη πρώτα απ' όλα την ε, λογιστική, τον ειδικό λογιστικό ε, έλεγχο για την περίοδο 13-20. Ε, είχαμε την πρώτη, τον πρώτο τριμερή διάλογο και στο άρθρο 4 έγινε, για το άρθρο 4 έγινε η περισσότερη συζήτηση ε, και ε, υπάρχει ε, μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τις διαφορές οι οποίες παραμένουν όσον αφορά το προτινόμενο εργαλείο. Ο δεύτερος τριμερής διάλογος θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου. Όσον αφορά όσον αφορά τον ε, ε, τριμερή διάλογο Μήφη, ε, έλεγε και εκεί η χώρα η πρώτη συνεδρία και εδώ ζητούμε περισσότερη διαφάνεια και συζητήθηκε το θέμα του reporting για τις τρίτες χώρες. Στις 6 Νοεμβρίου προβλέπεται και για το θέμα αυτό ο επόμενος διάλογος. Περνάμε τώρα... Α, στην ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Ελέγξτε αν έχετε όλοι τις κάρτες σας. So, we move on to the vote. Περνάμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία είναι μια δική μου έκθεση. Λοιπόν, να δούμε αν, λειτουργούν, ε, αν λειτουργεί το σύστημα, αν έχετε τις κάρτες σας. Κάντε, να κάνουμε λοιπόν μία πρώτη ψηφοφορία για να ελέγξουμε. So everyone vote? No, Ψήφισαν όλοι. Υπάρχει κάποια κάρτα που δεν λειτουργεί. Πέρασε τη ψηφοφορία. Ξεκινάμε λοιπόν Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση της κυρίας Κέι Συμβιβασμός ε, Α υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Ναι, η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 28. Πέρας της πληροφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός Β. Όχι. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός Β. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Α, έχει αποσυρθεί. Ωραία. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Έχει αποσυρθεί μου λέτε. Εντάξει, τροπολογία 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41-42 είναι ταυτόσιμες, δεν ψηφίζουμε. Άρα τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφοι 5-6 υπέρ. Κατά. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός C. Α, όχι, έκανα λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός C. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Σε ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός Δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία... Τροπολογία 52 τμήμα 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 τμήμα 2 έχει αποσυρθεί. Συμβιβασμός Ι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 με προφορική τροπολογία του εισηγητού, της εισηγητρίας μάλλον. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός Αι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφολογή, ε, συμβιβασμός J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 100. Votes, adopted. Εγκρίνεται. 18 ψήφοι υπέρ, 13 ψήφοι κατά. Σας ευχαριστώ πάντως. Ναι, αλλά έτσι πήρα και εγώ λίγο μια ανάσα. Συμβιβασμό εμ. υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Το αυθεντικό κείμενο, του πρωτότυπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογικό Αρχικό κείμενο. Θέλετε να ελέγξουμε την 110. Λοιπόν, εδώ στον κατάλογο έχουμε ότι πρέπει η, ψηφοφορία για τις 109 και 110 να γίνει ενιαία. Ωραία, μία ψηφοφορία για τις ε, τροπολογίες 109 και 110. On block λοιπόν 109 και 110. So we are both. Uh, Εντάξει, θα γίνει λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση για τις τροπολογίες 109 και 110 πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίνεται 15 ψήφοι υπέρ 14 κατά. Let's vote it separately then. There is no problem. We vote. Εντάξει, να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε. So, if there is uh, any concern, we vote separately. We vote. Ωραία, να ψηφίσουμε χωριστά. Ωραία. Την 109. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 109. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. 109. Πέρας της ψηφοφορίας. Και Απορρίπτεται. 4 ψήφοι υπέρ, 27 κατά. Ψηφίζουμε τώρα την 110. Άρχεται η ψηφοφορία. Και απορρίπτεται επίσης. 15 υπέρ, 16 κατά. Συγγνώμη, δεν είχα καταλάβει τι μου ζητούσατε. Προχωράμε λοιπόν. Τροπολογία, όχι μάλλον το αρχικό κείμενο, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 111 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης ε, αρχικό κείμενο για την θεολογική σκέψη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 4 και 5 μάλλον ψηφίζουμε από κοινού τις τροπολογίες 4 και 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο του εκτιμώντας 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο του εκτιμώντας 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο 5 και 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο αιτιολογική σκέψη α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε, το original text, ε, συγγνώμη, τροπολογία 12, ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση, δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Τροπολογία 12, δεύτερο τμήμα. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται 16 υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της αιτιολογικής σκέψης Δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο αιτιολογική σκέψη ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο αιτιολογικής σκέψης FG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο αιτιολογικών σκέψεων J και L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, ιδιολογική σκέψη M, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβασμός R, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, ιδιολογική σκέψη O, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 24 για την αιτιολογική σκέψη ΟΟΥ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε τώρα Α, θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 24 όχι ηλεκτρονική ξαναψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε τώρα το τροποποιημένο κείμενο ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται We close the vote adopted. Ψηφίζουμε. Και ψηφίζουμε τώρα για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 30 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια κυρία Σουίνμπερν. Επόμενη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την έκθεση Τρεμόζα για τον ανταγωνισμό για την πολιτική του ανταγωνισμού. Συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 13 υπέρ χωριστή ψηφοφορία μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται αλλά να τα επαληθεύσουμε το πρώτο μέρος τροπολογίας 13 άρχιτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να την επαληθεύσουμε Πέρας. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. 21 την προφορική τροπολογία του κ. Παλώνη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Να την επαληθεύσουμε την 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Με την πλειοψηφία. Ε, φαντάζομαι μόνο ο κύριος Λάμπερτς ψήφισε κατά. Τροπολογία 23 υπέρ. Η 22 έχει αποσυρθεί. Έτσι μας λένε. 23 υπέρ. 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές απορρί 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές δεκτή. 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή να επαληθεύσουμε την 52 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 54 χωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 59, 57, με συγχωρείτε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 63 υπέρ κατά αποχές 64 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Συμβαστική ε. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εν. Νι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 71. Απορρίπτονται. Εντάξει. 72 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική F υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 74 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 83 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Συμβαστική G σε δύο μέρη. μέρο πρώτο υπέρ. Κατά. αποχέ δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. αποχέ, δεκτή. Το μέρος δεύτερο της G. Ναι, το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία.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 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πρέπει να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο στην 93. Yes. Το αρχικό κείμενο, με συγχωρείτε, της ε, παραγράφου 11. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Σας ευχαριστώ, κύριε Γκοζές. 94 υπέρ κατά αποχές δεκτή 95 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 Α, το αρχικό κείμενο της παραγράφου 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 97 ε, και 98 υπέρ κατά αποχές δεκτές 100 ε, υπέρ Α, 99 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές δεκτή αρχικό κείμενο της παραγράφου 13 Α, όχι 100 υπέρ Κατά. Αποχές. Δεκτή. Να την επαληθεύσουμε όμως αν θέλετε. Πέρας. Εγκρίνεται. Βεβαίως. 101 υπέρ. Να με συγχωρείτε. Ε, καταπίπτει. Φάλος. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Αρχικό κείμενο, ναι. Ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αρχικό κείμενο, όχι 106, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 107, μέρος πρώτο, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 108 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές δεκτό 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή 114 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 116 να τα απολυθέσουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, μα νομίζω Μόνο οι βουλευτές μπορούν να ζητάνε επαλήθευση, έτσι, όχι το προσωπικό. Ε, υπενθυμίστε τους, σας παρακαλώ, το γεγονός. Σας ευχαριστώ. Ε, εγώ ακούω ένα τσεκ, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι βουλευτής ή όχι, αλλά σας παρακαλώ μόνο οι βουλευτές μπορούν να ζητάνε έλεγχο. Πέρας της ψηφοφορίας ε, εγκρίνεται. 117. Όχι καταπίπτει. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, Γκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή αρχικό κείμενο της ε, παραγράφου 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική I υπέρ κατά αποχές δεκτή 132 υπέρ κατά αποχές δεκτή 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο α όχι πρέπει να το ψήσουμε. 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή 136 και 137 υπέρ κατά αποχές δεκτές 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές δεκτή 143 υπέρ κατά αποχές δεκτή 144 υπέρ κατά αποχές δεκτή 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή 146 υπέρ κατά αποχές δεκτή 147 mm. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 και 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές δεκτή 153 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές δεκτή 159 υπέρ κατά αποχές δεκτή 155 υπέρ κατά αποχές δεκτή 160 υπέρ κατά αποχές δεκτή 157 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική K, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Απολογία 168, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική L. Ορίστε, παρακαλώ. Συμβαστική L, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές δεκτή 180 ταυτόσημη ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, έμπλ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή έμπλ 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 5 υπέρ σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ, κατά αποχές δεχτεί Να το επαληθεύσουμε. Πέρας. Δεκτή. Μέρος δεύτερο. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 6. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 6 μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έμπλ 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έμπλ 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έμπλ 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 14 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 15 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή έμπλ 16 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές δεκτή έμπλ 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή εκτιμώντας εκτιμώντας α υπέρ κατά με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 ε. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Υπέρ κατά αποχές δεκτός. Β. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. Ε, εκτιμώντας C ε, υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται εκτιμώντας δέλτα ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, εκτιμώντας ε υπέρ κατά αποχές δεκτό εκτιμώντας F υπέρ κατά αποχές δεκτό unblock οι αιτιολογικές αναφορές υπέρ κατά αποχές δεκτές συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές δεκτή ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το κείμενο όπως τροποποιήθηκε So we close the votes and 32 in favor. 32 υπέρ, ε, μία ψήφος κατά. Ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια στον κύριο Τρεμόσα. Περνάμε τώρα στα συνταγματικά προβλήματα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κυρίας Γκουλάρ. Συμβιβασμό Α υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Συμβιβασμό Β υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Συμβιβασμό Σ, Συμβιβασμό Σ υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Συμβιβασμός D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός E υπέρ. Κύριε Γκοζές, θα θέλετε επαλήθευση. Βεβαίως, τροπολογία 26, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ, 11 ψήφοι κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα το συμβιβασμό E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός H υπέρ κατά αποχές on block. Λοιπόν, από κοινού όλες, όλοι οι συμβιβασμοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται όλοι. Συμβιβασμός S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 καταπίπτει. Συμβιβασμός V. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός W μέχρι AJ. Θέλετε να ψηφίσουμε από unblock. Ε, Πολύ ωραία. Υπέρ. Παρατηρήσει εκτός μικροφώνου. Η, η, η τροπολογία 52 καταπίπτει. Ωραία και ψηφίζουμε λοιπόν τις, τους συμβασμούς από το W μέχρι το AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε λοιπόν από κοινού το τροποποιημένο, ε, ψηφίζουμε συγγνώμη το τροποποιημένο κείμενο. Πέρας της ψηφοφορίας. 26 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια κυρία Γκουλάρα επόμενο θέμα της μερησίας διάταξης. So we move on to the next item of the agenda. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα της μερικής διάταξης. Τροποποίηση του κανονισμού 99 κάθετος 2013 το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα για το 2013 με 17 του οποίου έχω την τιμή να είμαι εισηγητής. Please be Παρακαλώ ησυχάστε για να παρουσιάσω την έκθεσή μου στα ισπανικά. Όπως γνωρίζετε, η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής απαιτεί συγκρίσιμα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για οικονομική, και κοινωνική κατάσταση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και στις χώρες μεμονωμένα. Σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο τα στατιστικά αυτά στοιχεία είναι σημαντικά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι κάνει η Ευρώπη. Ο κανονισμός λοιπόν αυτός του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013-2017 που εγκρίθηκε στις 15 Ιανουαρίου φέτος με στόχο να καθορίσει ένα γενικότερο πλαίσιο για την ανάπτυξη και διάδοση των στατιστικών στοιχείων για το 2013 μέχρι και 2017 όπως είπα και προηγουμένως δύο φορές. Ο σχέδιο αυτό κανονισμού υποβλήθηκε από την Κομισιόν και ανέρχεται σε ύψος 292 εκατομμυρίων. Δεν υπήρξαν σοβαρές αντιρρήσεις κατά την εξέταση, αλλά παρόλα αυτά στις 13 Ιουνίου 2012 για το ΠολΔΙΠ και τους ιδίους πόρους το Κοινοβούλιο σε ψήφισμα του τόνισε ότι οι διατάξεις για τα πολιετή προγράμματα θα καταλήξουν όταν θα έχει υπάρξει συμφωνία για τα κονδύλια. 2013 en el programa estadístico europeo 2000. Επομένως και το στατιστικό αυτό πρόγραμμα 13 με 17 για τα κονδύλια του θα υποβληθεί σε αυτό το κανόνα. Είναι ένα τετραετές πρόγραμμα, το ξαναλέω για πέμπτη φορά, 2013 με 2017. Τετραετές, τέσσερα χρόνια δηλαδή. Και εμπίπτει στα πλαίσια του Πολδίπ μέχρι το 20. Η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα από το 2013 είναι 57 εκατομμύρια για το 7 μέχρι το 13, από το 7 μέχρι το 13 τα κοινωτικά κονδύλια. Μέχρι το 17 από το, θα είναι 234 εκατομμύρια. Και το πρόγραμμα που σας ανέφερα 7 φορές 13 με 17 θα παραμείνει ως έχει σε αυτά τα κονδύλια. Θα ήθελα τώρα να υποστηρίξουμε το, την πρόταση της Κομισιόν χωρίς τροποποίηση, χωρίς τροποποίηση, διότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Και ζητώ την υποστήριξη και των σκιωδών. Επίσης μου είπαν ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει την πρόταση και ο λόγος είναι ότι πρέπει να είμαστε <clears throat> αποτελεσματικοί. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή στην εικόνα και νομίζω ότι οι εκθέσεις για τα στατιστικά στοιχεία είναι από τις σημαντικότερες. Άρα καλό είναι να συνδυάζονται. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ και θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις, όσους τουλάχιστον είναι παρόντες. Κυρία Γκουλά, δεν έχω τίποτα να προσθέσω, λέει η κυρία Γουλάρ, σε διάφορες γλώσσες. Δεν νομίζω ότι είναι αμφιλεγόμενο το ζήτημα, επομένως μπορούμε απολύτως να σας στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκουλάρ. Οι πράσινοι μήπως έχουν κάποιο εκπρόσωπο, θέλει να μιλήσει κανείς, όχι, από τους συντηρητικούς, ο κύριος Σεπίνγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας στηρίξω πλήρως. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν ε, μακράν ναι, η συντομότερη συζήτηση. Η Κομισιόν πως θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς ε, να καλωσορίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ε, στήριξη. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ, είστε πάντα πολύ ανοιχτό στη συζήτηση τα τελευταία χρόνια και ελπίζω και με το νέο πρόγραμμα να συνεχιστεί αυτή η καλή κατάσταση. so have... Πάρα πολύ ωραία. Επομένως ε, δεν έχουμε κάποιον αγορητή που να θέλει το λόγο. Προθεσμία για, την υποβολή τροπολογιών 24 Οκτωβρίου, 24 Οκτωβρίου. Εάν υπάρξουν τροπολογίες θα ξανασυζητηθούν στις 19 Νοεμβρίου, θα ψηφίσουμε την ίδια μέρα και μετά θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του μηνός Ιανουαρίου. So we move on. We should move on. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή το υπαριθμό 8. Κανόνες για αποζημιώσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ένωσης. Ο εισηγητής ο κύριος Σβάμπ δεν είναι εδώ. Οπότε να βάλετε η συζήτηση μέχρι να έρθει ο κύριος ε, Σβάμπ, γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Διακόπτεται λοιπόν η συνεδρίαση και ελπίζουμε ο κύριος Σβάμπ να έρθει σύντομα.

Ah, so welcome, Mr. Swap. So we move on Ωραία λοιπόν να περάσουμε το, στο σημείο ε, στο σημείο 8 της ημερησίας διατάξεως κανόνες ε, η έκθεση του κυρίου Ανδρέα Σβάμπ κανόνες που διέπουν τις αγωγέ αποζημίωση βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσει των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σουάμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Πάμπλο, αγαπητή συνάδελφοι. Χαίρομαι για το ότι συζητάμε σήμερα για πρώτη φορά το σχέδιο έκθεσης για τις αποζημιώσεις για παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού και στο λίγο χρόνο που έχω θα ήθελα να παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της πρότασής μου και έτσι να συνεισφέρω ε, οι συζητήσεις που είχαμε διμερώς με τον κύριο Σάντσες Πρεσέντο από τους Σοσιαλδημοκράτες και τον κύριο Έπινγκ από τους Συντηρητικούς και ε, με την ε, κυρία Σόφι Νετφέλντ από τους Πράσινους ε, να συνοψιστούν. Νομίζω πως κάναμε μια θετική πρόταση και η Κομισιόν δηλαδή γιατί συμπεριέλαβε αυτά τα οποία έχει στήσει ήδη από το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή να διασφαλίσουμε οι άνθρωποι οι οποίοι πέσαν ζημίες ε, λόγω μονοπωλιακής συμπεριφοράς να αποζημιωθούν. Είναι βασική αρχή στην ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να υπάρχει αποκατάσταση των ζημιών. Γι' αυτό θεωρώ πως όλα πηγαίνουν, όλα αυτά είναι προς σωστή κατεύθυνση. πέρα δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πουθενά με την πρόταση αυτή περαιτέρω δυνατότητες. Απλά μπορούν να συνδυαστούν οι μέθοδοι που υπάρχουν στα κράτη-μέλη για να υπάρχει, αν θέλετε, η δυνατότητα ενός, να, να απευθυνθεί κάποιο σε μία υπηρεσία. Βεβαίως εδώ πέρα η αποζημιώσεις που δίνονται δεν έχουν ε, τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά ε, ο κύριος Φλόρεντς ε, είχε πει πως ελπίζει να επιτρέπεται, να συνεχίσουν να επιτρέπονται στην χώρα του. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, να μην δημιουργηθούν εδώ πέρα λάθος κίνητρα συνολικά. Η πρόταση της Κομισιόν προσανατολίζεται στο ότι οι ε, τροπολογίες ε, που έχουν κατατεθεί έχουν ως στόχο όταν υπάρχει ένας βασικός μάρτυρας ο οποίος δίνει πληροφορίες ε, να μην επιβαρύνεται ο ίδιος γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος επιβαρύνεται πάρα πολύ διατρέχει κίνδυνο με το να δώσει αυτές τις πληροφορίες και δεν είναι δυνατόν μετά να χρησιμοποιηθούν εναντίον του. Ο κίνδυνος λοιπόν το μείωσης αυτών των κινήτρων υπάρχει στις δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να και Μη και ε, Φλάιντερε καθώς ε, θεωρούσε το ΔΕΚ πως δεν υπήρχε επαρκής ε, νομική βάση, οπότε θα πρέπει οι συνθήκες υπό τις οποίες αποφασίζει ο δικαστής ε, το εάν θα πρέπει να υπάρξει αναζήτηση αυτών των πληροφοριών είναι οι σωστές. Η Κομισιόν εδώ πέρα προτείνει στο άρθρο 5 να υπάρχει ένα γενικό κάθεστος για τις εθνικές αρχές και τον δικαστή, δηλαδή να ελέγξει το εάν και κατά πόσον μπορούν να δημοσιευτούν έγγραφα που αφορούν τον ανταγωνισμό και βεβαίως φεύγουμε από αυτό το οποίο υπήρχε στο παρελθόν ότι ποτέ δεν θα έπρεπε να δημοσιευτούν. Για τα δε έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 6 δημιουργείται πλέον μια πλήρης νομική ασφάλεια αλλά έχουμε εδώ πέρα κάποια έγγραφα τα οποία έχουν μια ειδική μεταχείριση και άρα ο δικαστής μπορεί να οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως όλα τα υπόλοιπα μπορούν να δημοσιευτούν άφοβα. Αυτή η διάκριση ε, που είναι μόνο άσπρο μαύρο αν θέλετε δεν είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή και της ε, βεβαιότητας του δικαίου και αντιθέτως η Κομισιόν μπορεί πάντα να πει πως τα έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες Κομισιόν προστατεύονται ενώ όλα τα άλλα όχι. Εμείς λέμε να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση για όλα τα έγγραφα τα οποία εμπλέκονται σε διαδικασίες ε, ανταγωνισμού και να μην υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εγγράφων. Το ξεκαθαρίζει νομίζω και ο τίτλος του άρθρου. Ότι ισχύει δηλαδή για όλα τα είδη των έρευνων. Δεν θα αναφερθώ τώρα άλλο στα άρθρα 5 και 6 παρά το ότι είναι η ουσία της πρότασης. Ένα άλλο σημείο είναι τα συμφέροντα αφενός αυτών που ε, δημιούργησαν καρτέλ και το πώς θα συμβιβαστούν με τα συμφέροντα των ε, καταγγελόντων. Παίζει εδώ πέρα λοιπόν σημαντικό ρόλο η ε, συνολική ευθύνη η οποία υφίσταται. Η Κομισιόν λοιπόν έκανε μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Δηλαδή ο βασικός μάρτυρας ε, θα έχει προνομιακή μεταχείριση και στην επιμέτρηση της ποινή όχι μόνο όσον αφορά τα έγγραφα αλλά και όσον αφορά την ευθύνη του έναντι τρίτων. Ξέρω βεβαίως πως αυτό είναι επίμαχο, αλλά εξακολουθώ να θεωρώ πως ε, πάρα πολύ συχνά, πως ε, συχνά ο οικονομικά ε, ισχυρότερος είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί συνήθως σε αυτή τη διαδικασία επίσης. Όσον αφορά την ε, κοιλή και ελέγγυα ευθύνη, δεν θεωρούν πως θα πρέπει να επεκτείνεται, όπως σας είπα, στους βασικούς μάρτυρες. Η Κομισιόν ε, θεωρεί πως ε, εδώ πέρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να καταγγείλουν μια τέτοια κατάσταση νωρίτερα γιατί θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να αποδείξουν ποιες είναι οι ζημίες οι οποίες υφίστανται αυτό πράγματι είναι αναμφισβήτητο αλλά βεβαίως ε, το να έχει μετά πλεονέκτημα ως ε, ε, πιστοτής είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Επίσης, όσον αφορά υποθέσεις που γίνονται για τις πιθανές ζημίες, εγώ δεν είμαι υπέρ γιατί είναι κάτι το ρευστό το οποίο δεν μπορεί να αποδειχθεί με τρόπο άκλοντο και νομίζω πως ε, ε, εδώ πέρα όποιος το θέλει θα πρέπει βεβαίω να φέρει και το βάρος αποδείξεως και τον κίνδυνο να μην αποδειχθεί τελικά κάτι τέτοιο. Μίλησα με ε, ενός καταναλωτών, με επιχειρήσεις. Κανένας δεν είναι πολύ ικανοποιημένος. Ε, ίσως καταλήψουμε σε κάποιο συμβασμό. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω στο θέμα που θέτει η Κομισιόν στο άρθρο 17.3 για τις ε, νομικές διαδικασίες που προβλέπεται μπορεί να υπάρξει μια αποζημίωση, μια αποζημίωση στη βάση ε, εναλλακτικής επίλυσης ε, διαφορών, κάτι το οποίο βεβαίως είναι για εμάς ε, θετικό. Γι' αυτό όμως πρότεινα το 17.2α, όπου λέμε πώς θα πρέπει να δημιουργηθεί κάτι ανάλογο και στο πλαίσιο της Κομισιόν. Για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα όσων έχουν υποστεί ζημία με τρόπο οικονομικότερο. Νομίζω κάλυψα τα σημαντικότερα. Θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα στο χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για τι είναι η 5η Νοεμβρίου. Ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε 5η Δεκεμβρίου. Νομίζω πως τα άρθρα 5, 17 και 18 έχουμε το δικαίωμα της συναπόφασης με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε καιρός. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Σκιώδη Σάντσες Πασάρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ τον κύριο Σφάμπ για το έγγραφό του, καθώς και όλους τους άλλους κοιόδης για το, τη συνεργασία και τον διάλογο, κυρίως όμως τον εισηγητή. Δύο παρατηρήσεις. Εδώ μιλάμε για θέμα που στοχεύει στην διατήρηση του ρόλου μας ως, της δικαιοδοσίας μας ως αρμόδιας καθήλυν επιτροπής. επιτροπής. και όχι για καμία παρέμβαση στα εθνικά νομικά ή δικαστικά συστήματα. Ζητούμε απλώς περισσότερη αποτελεσματικότητα. Η Ένωση και η Κομισιόν δεν έχουν καμία πρόθεση να παραβιάσουν δικαιοδοσίες των χωρών μελών. με απλώς τη συνθήκη. Αυτή είναι ακριβώ η δικαιοδοσία της Επιτροπής μας και εμείς είμαστε οι αρμοδιότεροι να την προασπίσουμε. Είναι καθαρά θέμα ανταγωνισμού όπως είπαμε. που διαφέρει από τα οριζόντια θέματα και είναι ακριβώς δικαιοδοσία της Επιτροπής εικόνων. η διάδοση στοιχείων για τον ανταγωνισμό από τις αρμόδιες αρχές του ανταγωνισμού είναι ακριβώς αυτό το θέμα και υπάρχει και το θέμα των αποφάσεων των αρχών ανταγωνισμού. Γίνεται όταν μιλάμε για περιόδους εννοούμε φυσικά ιδιώτες. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικές προτάσεις για, δύο πραγματικότητα, για την ίδια πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα σύστημα ενθάρρυνσης αυτής της πολιτικής του ανταγωνισμού. Λοιπόν, όλα είναι θέμα αποτελεσματικότητας της πολιτικής ανταγωνισμού. όταν μιλάμε για ζημίες προς το περιβάλλον ή στα δικαιώματα των καταναλωτών, το θέμα σχετίζεται και με αυτό. Εμείς λοιπόν είμαστε οι αρμόδιοι και το λέει ρητά ο κύριος Σουβάμ, αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανταγωνισμού. Αλλιώς δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης αυτή η πρωτοβουλία. Αυτό ήταν το ένα το οποίο θα ήθελα να απευθύνω και προς τον εισηγητή και προς την πρόεδρό μας. Τώρα το 2. Πρέπει νομίζω να δεχτούμε να συμφωνήσουμε τις μεγάλες κατευθυντήρες γραμμές της πολιτικής μας. <clears throat> δηλαδή να, βρεθούμε, να βρεθούν λύσεις. Αφού υπάρχει κάποια πολιτική ισορροπία, κάποια πολιτική συμφωνία, μετά πρέπει να δούμε τα πρακτικά τις πρακτικές λεπτομέρειες. Οι συλλογικές προσφυγές εδώ δεν αναφέρονται και ίσως αυτό να είναι μια έλλειψη. Πρέπει κάτι να πούμε και γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να τονίσω τα εξής. Όταν μιλάμε για πρόσβαση σε αποδείξεις, αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχει μια σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήδη, provocar la indefensión. Y por lo tanto, no hay ningún derecho absoluto. Todos los derechos deben facilitar el reconocimiento del derecho a la defensa y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 δεν είναι λογικό να τους θέτουμε τέτοιο βάρος σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ούτε θέλουμε να χρησιμοποιούνται οι μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις ως μοχλός κατά τον καρτέλ. Κάτι άλλο πολύ λογικό είναι η σχέση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Είναι δύο διαφορετικοί τομείς. και πρέπει να ενθαρρύνουμε την συνέργεια μεταξύ τους με συνέπεια προς τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι δημόσιες αρχές. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ενιαίο σύστημα κυρώσεων να υπάρχει κάποια συσχετισμός μεταξύ, δηλαδή αναλογία μεταξύ της ζημίας και της κύρωσης. Αλλά ούτε θέλουμε να επιβαρύνουμε τώρα την Κομισιόν πολύ με τα ιδιωτικά. Δεν είναι η δουλειά τους. Εκείνοι ασχολούνται περισσότερο με τα δημόσια θέματα και δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε περισσότερο την διοίκηση με την αξιολόγηση των ιδιωτικών ζημιών γιατί αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικίνητρο στην πολιτική ανταγωνισμού. Να το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Για τα χρονοδιαγράμματα τώρα στον Ισπανικό νόμο, στην Ισπανική νομοθεσία προβλέπεται ένας χρόνος εδώ πέντε. Και δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε την περίοδο των περιορισμών για τον ιδιωτικό τομέα τις ιδιωτικές ζημίες με ό,τι ισχύει στο δημόσιο τομέα. Τα θύματα δηλαδή κάποιου καρτέλ δεν μπορεί να αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους και τα αράλληλα να λέμε ότι «Α, ναι, αλλά πέρασε η διορία». Πρέπει η περίοδος του περιορισμού να είναι λογική. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε χρόνια. Και άμα περάσουν τα πέντε χρόνια, άμα περάσουν, να υπάρχει και κάποια άλλη διορία για να μπορεί κανείς να προσφύγει. Για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανταγωνισμού δεν αναφέρομαι σε συλλογικές προσφυγές, αλλά στην αποζημίωση μικρότερων ζημίων. και αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι πολύ δύσκολο να ζητήσει κανείς αποζημίωση για μικρές ζημίες, αλλά καμιά φορά ορισμένες εταιρείες προσφεύγουν και σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει και γι' αυτό να προβλεφθεί κάποια διαδικασία. Για να μην υπάρχει ατιμορρησία. Όπως γίνεται σε άλλους νομικούς τομείς. Αποφεύγοντας πάντοτε βέβαια τους υπερβολές των ΗΠΑ. Αυτά είχα να σας πω. Είναι σε καλά χέρια η έκθεση, έχει εμπειρία ο κύριος Βάμπη αυτά τα θέματα και μέχρι τώρα συμφωνήσαμε σε πολλά μεταξύ μας και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και γενικότερα πριν λήξει αυτή η θητεία. Ευχαριστώ. Ο Ανδρέας Σβάμπ πρέπει να πάει να ψηφίσει στην Ίμκο. Γι' αυτό έφυγε. Το γραφείο του όμως οι εκπρόσωποι του γραφείου του θα σημειώσουν ό,τι έχετε να πείτε. Κυρία Γκουλάρ, εξ ονόματος της Σοφίας. Όχι, δεν έχω τίποτα να πω εξ ονόματος της Σοφίας, έχω να πω όμως εξ ονόματός μου. Ε, ο κύριος Βαμ μπορεί να φύγει, να ψηφίσει με την ησυχία του. Δεν έχω να πω τίποτα. Λοιπόν, θα πρέπει να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αντωνίου Πετσέρο γιατί είναι ο ε, πρεσβύτερος από τους παριστάμενους και πρέπει να του δώσω τη θέση μου. Θα προεδρεύσει μέχρι το τέλος της συνεδρίας. ελπίζω ότι μέχρι να τελειώσω τη δικιά μου παρέμβαση θα έχει μείνει και κανένας βουλευτής στην αίθουσα. Κρίμα που φεύγει ο κύριος Βαμπ. Γιατί θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τον ευχαριστήσω ε, για την εργασία που έχει εκπονήσει μέχρι τώρα. Αλλά και δεύτερο, είμαστε κάπως επικριτικοί απέναντι στην εργασία του κυρίου Σβάμπ, γιατί βλέπει, βλέποντας κανείς ε, την ε, εργασία της Κομισιόν, έχει την αίσθηση ότι πρέπει να την τονώσει, να την ενδυναμώσει. Και δεν την ενισχύει καθόλου την πρόταση της Κομισιόν ο κύριος Σβάμ. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, φτάσουμε σε κάποια συμφωνία αρκετά γρήγορα, αλλά δεν θα είναι και εύκολα τα πράγματα. Γιατί κατά τη δικιά μας άποψη το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν θέλουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση η οποία τελικά είναι επωφελής μόνο για τις επιχειρήσεις και όχι για τους καταναλωτές. Θέλουμε ε, μια καλή ανοιχτή αγορά σε καλές συνθήκες ανταγωνισμού χωρίς ε, ε, ζημίες και άσχημες καταστάσεις για τους καταναλωτές. Η κατάσταση σήμερα είναι προβληματική. Πολύ συχνά, υπερβολικά συχνά μάλλον, ε, χρησιμοποιούνται από πλευρά των επιχειρήσεων ε, διάφορες ε, επιχειρηματολογίες για την μη αποζημίωση και φτάνουμε όσο γίνεται περισσότερες, όλο και περισσότερο στο δικαστήριο. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης, ικανοποίησης δηλαδή αυτών των αγωγών αποζημίωσης από μεμονωμένους πολίτες. γιατί είμαστε πάντα πάρα πολύ προφυλακτικοί, ε, πάρα πολύ προσεκτικοί και το πρώτο μέλημα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων της βιομηχανίας. Όμως, ο καθένας μεμονωμένος καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποζημιωθεί σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημία. Θέλουμε λοιπόν ενίσχυση του κανονισμού. Και μία από τις συζητήσεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ε, πολύ, είναι η έλλειψη συλλογικής προσφυγής. Καταλαβαίνω ότι από πλευράς της Κομισιόν θα ήθελαν πριν τις εκλογές να έχει κλείσει το θέμα αυτό. Ίσως φοβούνται να ε, ξανανοίξουν τη συζήτηση ε, της ε, συλλογικής προσφυγής. Αλλά χωρίς συλλογική προσφυγή για αυτούς τους κανόνες είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Θα ξεκινήσει λοιπόν ελπίζω η συζήτηση, το περιμένω και ελπίζω να κλείσει και με σωστό τρόπο. Δεύτερον, πρόσβαση σε στοιχεία. Και εδώ έχουμε προβληματική διαχείριση του θέματος. Υπάρχει περιορισμός υπερβασιμότητα σε ορισμένα έγγραφα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε, μάλλον υπάρχει ε, υπάρχει μια διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την, την προσβασιμότητα των εγγράφων ε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να έχει κανείς τα έγγραφα τα οποία χρειάζεται έτσι ώστε να αποδείξει την ζημία που έχει υποστεί. Γι' αυτό λοιπόν Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διατύπωσή μας όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, γιατί πολλές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να ε, περιγράψουν τον νόμο. Ε, δεύτερον, ο ρόλος που έχουν ή πρέπει να έχουν οι αρχές του ανταγωνισμού έτσι ώστε να ε, μην ε, ε, υπάρξουν στο μέλλον υπερβολικές πολλές περιπτώσεις αγωγών αποζημίωσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει οι διάφορες αρχές να, είναι, να έχουν συμπληρωματική δράση. Εν συνόψη λοιπόν, στις δικές μας τροπολογίες θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην, στον ρόλο που παίζουν οι παραβιάσεις ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις, θα πούμε ότι η έλλειψη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ε, οφείλεται σε ελλειπή πληροφόρηση και ελλειπή δυνατότητα ε, ε, αίτησης αποζημίωσης και αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί και να λυθεί. Επίσης δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε απ' έξω το θέμα των συλλογικών προσφορών. Οπωσδήποτε θα πρέπει να το συζητήσουμε και στα πλαίσια αυτού του φακέλου. Περιμένω και τη συζήτηση βεβαίως με τον κύριο Σβάμπ. Ε, πρέπει... Έχουμε ακόμα διαφορετικές απόψεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε για να βρούμε κοινά σημεία ε, και σημεία επαφής, αλλά ελπίζω να μπορούμε να το καταφέρουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Έπινγκ έχει το λόγο από την ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ λιγόλογο θα είμαι σήμερα. Η μεγαλύτερη ομάδα νομίζω ότι απουσιάζει παντελώς ε, σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα των συντηρητικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στηρίζει τις ε, αγωγές αποζημίωσης και ελπίζουμε ότι ο κανονισμός θα εγκριθεί πριν το τέλος της δικιάς μας θητείας. Ο κύριος Σουάμπ δεν είναι εδώ, αλλά ελπίζω ότι τα μέλη του γραφείου του θα ε, του μεταφέρουν τα συγχαρητήριά μου. Ε, το θέμα των, ε, αστικών δικαστηρίων αγωγών αποζημίωσης με βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνο. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι και τα, και τα προγράμματα προστασίας των μαρτύρων και η παροχή κάποιων αντισταθμιστικών και τα προγράμματα επίοικια που προβλέπονται για τους μάρτυρες θα πρέπει να διατηρηθούν. Ε, επίσης ε, υπάρχουν και κάποια μικροσημεία, λεπτομέρειες ε, στην έκθεση που μπορώ να τα ρυθμίσω υποβάλλοντας τροπολογίες και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις σε ένα πνεύμα συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Έπινγκ. Δεν έχει δει κάποιος άλλος τον λόγο, οπότε θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στην Κομισιόν που μας θυμάμαι την παρουσία της ε, να τοποθετηθεί αν θέλει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας τα λόγια του κύριου Αλμούνια, ο οποίος ήρθε κατευθείαν στην Επιτροπή σας μετά την υιοθέτηση της πρότασης αυτής στο Ιούνιο, λέγοντα πως χαίρεται ιδιαίτερα που έχουμε αυτόν τον, το πρώτο φάκελο νομοθετικό περί ανταγωνισμού στο Κοινοβούλιο και θα αναλάβει το Κοινοβούλιο τον ρόλο του ως συνομοθέτης. Επίσης είμαι ικανοποιημένος ακούγοντας ε, την αναγνώριση του εισηγητού και των λοιπόν βουλευτών ε, για το ότι η Κομισιόν έλαβε υπόψη τα πολλά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν ήταν πάρα πολύ προσεκτική και προσπάθησε να ευθυγραμμιστεί με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου έχοντας δύο στόχους. Δηλαδή, να ενισχύσει την επιβολή από ιδιώτες ως ε, συμπλήρωμα της δημόσιας επιβολής και να διασφαλίσουμε τη συνύπαρξή τους χωρίς ε, μία να κινδυνεύει από την άλλη. Και ακούγοντας τις παρεμβάσεις των βουλευτών ότι συμφωνούν με αυτούς τους στόχους, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα. Θα τα λοιπά, κύριε Πρόεδρε, η Κομισιόν είναι πάντα στην διάθεσή σας για να διευκρινίσει την πρότασή της όπου αυτό χρειάζεται και ελπίζω να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην διαδικασία και εδώ στο Κοινοβούλιο και μετά στη συνεργασία με το Συμβούλιο. Η Κομισιόν θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα σέβεται τους δύο αυτούς αρχικούς στόχους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος τον λόγο. Οπότε, θα να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες, όπως είπε ο κ. Φαμπ, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Μετά θα εξεταστούν στις 25 Νοεμβρίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 5 Δεκεμβρίου. Έτσι έχει το πρόγραμμα για το θέμα αυτό. Έχουμε τώρα το σημείο 9 στην διάταξη. Είναι που έχουμε λίγο χρόνο. Προχωράμε γιατί είναι εδώ η συγητής. Έχουμε την ετήσια έκθεση 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο κύριος Τάις Μπέρμαν είναι εδώ, σοσιαλιστής και εάν δεν τον πειράζει τότε θα δώσω τον λόγο στον κύριο Μπέρμαν για να κάνει μια εισαγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί την θεωρώ ως βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη δική της οικονομία αλλά και για τη βελτίωση της οικονομίας των αναπτυσσομένων χωρών. Ως μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό το ρόλο του ΕΤΕ. Τώρα, για την έκθεση του 12. Φυσικά δεχόμαστε ότι είναι βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της κρίσης η ΕΤΕ και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μεγαλύτερη αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και την οικονομία της γνώσης και η διπλασιασμός του κεφαλαίου της με 10 δισεκατομμύρια ήταν σωστό, σωστή κίνηση. Αντίθετα όμως από αυτήν. Το επίπεδο υπογραφών είναι, δεν είναι ικανοποιητικό. Ο αριθμός των προγραμμάτων δηλαδή που μπορεί να χρηματοδοτήσει η ΕΤΕ ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερους από τους πόρους της πιο ενεργά για να μπορεί να αυξήσει τη δανειοδοτική της δραστηριότητα. δέχομαι τα πιλωτικά ομόλογα που προβλέπονται εδώ και ελπίζω να αυξηθεί η χρήση τους αν και η κυβέρνηση της χώρας μου δεν είναι πολύ ικανοποιημένη από αυτό. Μην γελάτε παρακαλώ. Είναι εδώ οι αντιπολιτευόμενοι στην Ολλανδία τέλος πάντων. Αυτές οι δραστηριότητες βέβαια πρέπει να γίνονται με αξιόπιστους εταίρους χωρίς τη χρησιμοποίηση φορολογικών παραδείσων κλπ. και με κανόνες διαφάνειας κλπ. Όσο για τη διαφάνεια η ΕΤΕ έχει μία ειδική διεύθυνση ελέγχου σε συνεργασία και με την Παγκόσμια Τράπεζα έτσι ώστε να γίνεται σεβαστή η αρχή της due diligence. Δεν βλέπουμε να, γίνονται, να υπάρχει όμως και πολύ μεγάλη διαφάνεια γενικά στις δραστηριότητες αυτής της Γενικής Διεύθυνσης για την επιμέλεια. Θα θέλαμε να υπάρχει έκθεση αναφορά ετήσια και για αυτήν. Επίσης, η διεύθυνση αυτή της ΕΤΕ δεν έχει μεγάλη πρόσβαση στις, στα πρακτικά των εσωτερικών συνεδριάσεων της ΕΤΕ. Αυτό μου φαίνεται πολύ περίεργο γιατί η διεύθυνση αυτή η μόρφωσης πρέπει να έχει πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων που είναι σημαντικές για την ποιότητα των δραστηριοτήτων της. Και ζητώ από την ΕΤΕ να δώσει αυτή την πρόσβαση στην διεύθυνση συμμορφώσεων. Βέβαια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και έξω από αυτήν είναι ουσιώδεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες στον κόσμο και στην Ευρώπη και η υποστήριξη από την ΕΤΕ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι Υπάρχει αλλά είναι άγνωστη γενικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Εχθές είδα κάτι εργοδότες από την Ολλανδία που δεν ήξεραν καν ότι υπήρχε δυνατότητα να συνεργαστούν με την ΕΤΕ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό εδώ η γνωμοδότηση ζητάει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες συνεργασίας της ΕΤΕ με ιδιωτικές τράπεζες για να γίνουν γνωστές οι δυνατότητες αυτές που δίνονται δανειοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ίσως έτσι να μειωθεί και το πρόβλημα της έλλειψης βιώσιμων προγραμμάτων που υποβάλλονται στην ΕΤΕ. Να, αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κύριο Κύριος τώρα. Α, όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Μου λένε ότι ζήτησε το λόγο εξονόματος της ομάδας της η συνάδελφός μας κυρία Γουλάρ. Ευχαριστώ. Εδώ αντικαθιστώ τον κύριο Σκυλακάκη που ήθελε να δηλώσει το εξής. Δύο πράγματα. Ας τα πω αγγλικά, ας πω αγγλικά. Ζητάει από την ΕΤΕ ετήσια να κάνει έκθεση για τις δανειοδοτήσεις της με συνδυασμένα στοιχεία για τις επιστροφές και που δίνει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υπάρχει έτσι κτλ. Ο Θεόδωρος λοιπόν θα ήθελε λίγο παρα περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πολύ συγκεκριμένο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συμφωνώ και εγώ. Δεύτερον, θα ήθελε να θέσει το θέμα ποια, ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο εάν στην περίπτωση που οι τοπικές τράπεζες δεν εφαρμόζουν τα προγράμματα λόγω έλλειψης ρευστού. Μπορούμε να προτείνουμε κάτι γι' αυτό γιατί είναι και αυτό σημαντικό θέμα για τον Νότο ιδιαίτερα. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι σημαντικό για όλες τις χώρες μέλη. Ευχαριστούμε Σιλβί. Και τώρα ο κύριος Έπινγκ. Ορίστε κύριε μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να στηρίξω τα περισσότερα από τα σημεία που ανέφερε ο εισηγητής, κυρίως δε όταν καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει την δανειοδότηση που θα βοηθήσει την δημιουργία θέσεων εργασίας, άρα να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα, τα ομόλογα έργου ε, θα πρέπει ε, να ε, υπάρχει τακτική αναθεώρηση έτσι ώστε να χρηματοδοτούνται εναλλακτικά ε, προγράμματα για τις ε, υποδομές κλπ. Επίσης να επιδειχθεί η due diligence έτσι ώστε να μην υπάρξει φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή ε, η, τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεργάζεται με τις αναπτυξιακές τράπεζες. Τέλος, να επιμείνουμε ε, στην ε, ε, αναλυτική έκθεση των δραστηριοτήτων κυρίως που αφορούν την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να γίνεται λοιπόν τακτική αναφορά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριε Επίνγκ. Ο κύριος έκων των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ε, ε, Τάις, εννοώ τον κύριο Μπέρμαν, ε, για αυτήν την γνωμοδότηση η οποία είναι ενδιαφέρουσα γιατί την βρίσκουν καλή και η ECR και η συντηρητική και η πράσινη. Κάτι σαθρό υπάρχει εδώ μάλλον, δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τα αστεία. Ε, ξέρετε, είναι αυτή η Βέλγο-Ολλανδική συμμαχία εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ε, κρίμα που το ΕΛΚ δεν είναι παρόν για να σχολιάσει. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου της κυρίας Γκουλάρ. Ναι, ακριβώς και εγώ θα έλεγα αυτό. Οποτεδήποτε μιλάμε για πειθαρχία και οποτεδήποτε μιλάμε για ανάπτυξη, φαίνεται ότι το ΕΛΚ λείπει, εν πάση περιπτώσει. Είναι καλό που στη γραμμοδότησή σας εστιάζετε την προσοχή σα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ θετικό. Να προσθέσουμε όμως και δύο-τρία πραγματάκια θα ε, θυμηθούμε και μία, μάλλον εδώ καλό θα ήταν να γίνει αναφορά ε, και σε ε, μία έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη των πόρων όσον αφορά τώρα την συγχρηματοδότηση προγραμμάτων είναι καλό που το αναφέρετε αλλά ε, είναι σωστό να υποστηρίξουμε ακόμα μεγαλύτερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, ε, στις υποδομές ενέργειας, κυρίως σε μη συγγνώμη, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. και όλα αυτά τα ζητήματα της ανάπτυξης που είναι σημαντικά και για την Νότια Ευρώπη. Εδώ θα προσθέσουμε μερικά πράγματα. Αλλά σε γενικές γραμμές έχω την αίσθηση ότι μπορεί αυτή η γνωμοδότηση να, γίνει, να είναι πάρα πολύ ε, ισχυρή. Και γι' αυτό λοιπόν ε, σε ευχαριστώ Τάις ε, για όσα έκανες μέχρι τώρα και θέλω να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Και Κρίμα που θα πρέπει να κάνω εκστρατεία εναντίον σου γιατί θα είσαι επικεφαλής της λίστας των σοσιαλιστών. Πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί. Ωραία λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, είναι γεγονός ότι προχωράμε πολύ γρήγορα στην ημερήσια διάταξη. Και αν θέλει ο κύριος Λάγκεν μπορεί να πάρει το λόγο. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα που έχει να μιλήσει. Δεν πειράζει. Θέλει ο κύριος Μπέρμαν να κάνει κάποια επιπλέον σχόλια μετά από τις ε, παρεμβάσεις που άκουσε ο κύριος Μπέργμαν. Μπέρμαν, ναι, ευχαριστώ. Σημειώνω με ευχαρίστηση όλες τις, ε, όλα τις παρατηρήσεις και τα σχόλια νομίζω ότι είναι σημαντικό που έχουμε μια σε γενικές γραμμές παρόμοια ανάλυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, την οποία θέλουμε να είναι αντικυκλική ε, και αποτελεσματική. Και είναι πολύ καλό που συμφωνούν ε, τα μέλη της Επιτροπής. Συμφωνώ, Σιλβί, ότι χρειάζεται αναφορά των αποτελεσμάτων όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά το αναφέρω στην έκθεση εδώ, γιατί ζητώ να γίνει αναφορά δικτών απόδοσης. Για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεσματικά πρέπει να ξέρουμε τι λειτουργεί καλά, τι έχει αποτελέσματα και τι όχι. Κύριε Έπινγκ, ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι θα πρέπει σε τακτικά διαστήματα να αναθεωρούμε ε, τα αποτελέσματα των project bonds, των ομολόγων έργων. Δεν μπορεί να τα ρίξουμε στη θάλασσα και να ε, κολυμπήσουν μόνα τους υπογραμμίζεται την ανάγκη αναφορά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Άλλωστε, αυτό είναι και το τελευταίο σημείο τη ε, έκθεση, ε, όπου λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να ενημερώνει συστηματικά για την πρόοδο που συντελείται σε σχέση με τι προηγούμενε συστάσει του Κοινοβουλίου. Και μπα σε ευχαριστώ βεβαίω. Δεν θα είμαι μαζί σου ε, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα εδώ είμαι, δεν χρειάζεται να μου βγάζει τον επικίδιο πριν φύγω. I have to Νομίζω ότι πρώτον σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μου είπες. Ε, θεώρησα ότι έπρεπε να μείνει λιγόλογη και σύντομη αυτή η ε, γνωμοδότηση. βεβαίως στο πέρασμα προς την, στη μετάβαση προς την αηφόρο οικονομία, ναι, μπορεί να γίνει εργαλείο σωστό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά δεν πρέπει να τη βαρύνουμε και πάρα πολύ. Κλιματική αλλαγή, ναι, φυσικά, φυσικά. Ε, ε, είναι απαραίτητη η μετάβαση προς την αηφόρο οικονομία και προς την στήριξη μη ε, συμβατικών μορφών ενέργειας. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται και θα συμπεριληφθούν και περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την τελική σας παρέμβαση. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το σημείο 9. Να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Για την γνωμοδότηση αυτή λοιπόν, 6 ε, Νοεμβρίου εκπνέει η, υποβολή, η προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών. 25 Νοεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 16 Δεκεμβρίου. Και η Επιτροπή ελέγχου του προπολογισμού θα συζητήσει το θέμα αυτό τον Ιανουάριο ε, και ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου για να συζητήσουμε το θέμα αυτό στην Σύνοδο της Ολομελίας του Φεβρουαρίου επαναλαμβάνω. Λοιπόν, έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα, αλλά από τη στιγμή που έχουμε εδώ τον ε, εισηγητή κύριο Κούτας, νομίζω ότι δεν ε, υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να συνεχίσουμε τη σε διάταξη και να ασχοληθούμε με το δικό του ζήτημα. Το θέμα του λοιπόν είναι η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα. Η είναι ο κύριο Ζόρζο Σαμπίν Κούτας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και του δίνω το λόγο αμέσως. Ευχαριστώ Αντολίνα. Για τα πρακτικά να υπενθυμίσω ότι για το θέμα αυτό η Κομισιόν προτείνει να διευρυνθεί η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ε, στα πλαίσια της ενίσχυσης ε, του, ε, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες θα αφορούν τις μετοχές, την κατανομή κερδών στους μετόχους κτλ. όλα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η μετάβαση σε μια καλύτερη ε, αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος που προέδρασε Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Επίσης, ε, ε, θα συνεχιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ, όπως έχει ήδη αποφασιστεί προτείνω στο κείμενο κάποια σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Είναι η προστασία των δεδομένων πρώτα απ' όλα, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ε, συμμόρφωση με τα όσα προβλέπει ο νόμος ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, υπάρχουν επίσης τα άρθρα 16 και 25 στην, οδηγία, στην αντίστοιχη οδηγία του Συμβουλίου αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ε, εξελίξεις όσον αφορά το διαδίκτυο θα πρέπει αυτές ε, οι διατάξεις τα στα άρθρα αυτά να ενδυναμωθούν. Επίσης ε, θα πρέπει η Κομισιόν να είναι πολύ προσεκτική όσον αφορά τις, την διαπραγμάτευση περαιτέρω πληροφοριών διμερών συμφωνιών με άλλες χώρες ε, για την ε, αυτό με την ανταλλαγή πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οι συμφωνίες οι οποίες έχουν ήδη διαπραγματευτεί δεν ε, υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξουν για να υλοποιηθεί σωστά η οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, όλα τα οικονομικά και τεχνολογικά, όλες οι οικονομικές και τεχνολογικές δυνατότητες οι οποίες παρέχονται. Οι κυρώσεις Η οδηγία αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή μεταξύ εθνικών αρχών. Ε, παρόλα αυτά θα πρέπει να ε, ε, προβλέπεται δεσμευτική να προβλέπονται δεσμευτικές κυρώσεις όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι. Οφείλω να συμφωνήσω ότι κάποιες από τις τροπολογίες βελτιώνουν το κείμενο, κυρίως δε συμφωνώ με τις τροπολογίες Uh, Πολλών συναδέλφων όπως ε, Μπασέσκου, Κάρεντς κλπ. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, ε, τροπολογίες οι οποίες απαλήφουν κάποια τμήματα του αρχικού κειμένου της Κομισιόν ή μειώνουν τον αριθμό των κατηγοριών ή θεμάτων που θα αφορούν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βρω κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες για τις αιτιολογίες σκέψης 1, 3 και 5. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ε, παράγραφοι οι οποίες είναι νέοι, νέες ε, και εδώ υπάρχει με μικρότερο περιθώριο των ε, για, για συμβιβασμούς. Ε, βεβαίως, ε, εάν οι συνάδελφοί μου θέλουν να συναντηθούμε, να, να κανονίσουμε συνάντηση με τους σχεδόν μπορούμε να το κάνουμε στο Στρασβούργο. Ε, μπορώ τώρα να ακούσω τα σχόλια ε, όλων των συναδέλφων και πριν τελειώσω να ευχαριστήσω και τον Μάρκο για την συνεργασία του. Ευχαριστώ. George. Ο κύριος Ζήτρας δεν είναι εδώ, αλλά ζήτησε ο λόγο η κυρία Γεροβιάσκα. Α, όχι, όχι. Δεν είναι εδώ οι ενδιαφερόμενοι. Θα δώσουμε το λόγο λοιπόν στην κυρία Γκουλάρη, η οποία ε, θα παρέμβει ο ξενόματος της ομάδας Άλντε. Ναι, βλέπετε ότι παίζω ολόκληρη ορχήστρα μόνη μου, λοιπόν. Δυστυχώς ε, δεν είναι εδώ ενδιαφερόμενος και μου ζήτησε να του αναφέρω τα Ε, Θεωρεί πολύ σημαντικό η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών να επεκταθεί για να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διμερείς συμφωνίες που έχουμε συνάψει με τα Συνωμένα Πολιτείας. Το λέει και στις τροπολογίες του. Βέβαια πρέπει να σεβόμαστε την ακαιρεότητα του κάθε προσώπου και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα προσωπικά του δεδομένα και γι' αυτό εξ ονόματος των φιλελευθερών και αυτό ήθελα να σας πω θα ζητήσουμε γνωμοδότηση από τον Ευρωπαίο ε, υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ελπίζουμε να μας απαντήσει σύντομα και βέβαια ο κύριος Σμιτ είναι στη διάθεσή σας για συμβιβασμούς. Muchas gracias, Silvi. Κούτας Όχι. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλε. Ξέρω για την ε, πρωτοβουλία του, για τη σύνταξη αυτής της επιστολής φοβάμαι πως ε, καθυστερήσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να επιταχύνουμε λίγο την διαδικασία αλλά βεβαίως ε, είμαι περίεργος για το τι θα γίνει αλλά να είστε σίγουροι πως όλα τα ζητήματα προστασίας των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικά έχουν καλυφθεί πάρα πολύ καλά Μόλις τροποποιήσαμε επίσης την αρχική οδηγία που περιέχει αρκετά τέτοια στοιχεία. Δεν αλλάζουμε τίποτα λοιπόν ως προς αυτό. Νομίζω... Κοιτάξτε, ο βοηθός του Όλε μου είπε κάτι Όλοι ήρθε σε επαφή μαζί τους και υποσχέθηκαν κάτι για την επόμενη εβδομάδα, οπότε δεν υπάρχει καθυστέρηση. Συμφωνώ μαζί σας πλήρως, δεν έχουμε σκοπό να καθυστερήσουμε τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ήρθε ο κύριος Μπέσε από τους Πράσινους, ο οποίος είχε ζητήσει να μιλήσει και η κυρία Γεσλοβέσκα επίσης μπήκε στην αίθουσα. Οπότε αν σας πειράζει θα τους δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Κύριος Μπέσε. Ναι, ε, είμαι εδώ εκπροσωπώντας τον συνάδελφο Ρουίς ο οποίος σας ζητεί συγγνώμη, δεν είναι δυνατόν να παραστεί. Είμαι λοιπόν εδώ ε, για να ευχαριστήσω εκ μέρους του τον εισηγητή. Το άλλο μου σχόλιο από την ομάδα των Πρασίνων θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή έχει πάρει τη σωστή κατεύθυνση, όπως ήθιστε να λέμε, κυρίως όσον αφορά τα θετικά ακόλουθα στοιχεία. Την διεύρυνση του πεδίου φορολόγησης εκτός προσωπικού, των στοιχείων προσωπικού πλουτισμού. Δηλαδή ότι οι διαπραγματεύσει με τις τρίτες χώρες θα πρέπει να είναι πιο ε, έντονες, ε, να είναι πιο ισχυρές και να είναι πιο ε, σαφής η εντολή και πιο περιεκτική. Μία παρατήρηση όμως, εδώ υπάρχει απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή και το δικό θεσμικό όργανο και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα να καθαρίσει πρώτα τα του οίκου της γιατί έχουμε την Αυστρία και το Λουξεμβούργο ε, που εξακολουθούν να είναι προσκολλημένες ε, ε, το τραπεζικό απόρριτο. Eh, ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε, η κυρία Γιαραβέσκα. Dziękuję Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εκπροσωπώ τον κύριο Μέτρας ε, που δυστυχώς οψιάζει. Θα ήθελα να σας πω τη δική του άποψη λοιπόν Υποθέτω ότι μπορώ να προσωπήσω τον συνάδελφο, έτσι. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, κύριε και κύριοι, με συγχωρείτε για την απουσία μου σήμερα, αλλά είχα κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ε, Βρίσκομαι σε συνεδρίαση του προεδρίου του ΕΛΚ, ε, εκτός ε, Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου. Το είχα πει πολλές φορές όταν ξεκινήσαμε να εξετάζουμε αυτή την οδηγία πως πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ευρώπη προς σωστή κατεύθυνση. Επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής της ανταλλαγής πληροφοριών σε νέου είδους κεφαλαία και εισοδήματα, όπως παραδείγματο χάρη μερίσματα, μετοχές κτλ. Σημαντικό αυτό για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές. Πρέπει όμως να υπάρξει κάποια βελτίωση και χαιρούμε για το ότι υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που συμφωνούν. Θα ήθελα να επισημάνω το ότι δεν ναι, ναι, έθιξα μόνο εγώ το ζήτημα κάποιων ανακριβιών ή έλλειψης νομικών ορισμών, ορισμένων κατηγοριών εισοδήματος και κεφαλαίου. Το θέμα αυτό ετέθη και από τον Όλε Σμιτ, ο οποίος είπε πως ε, αν δεν είναι ακριβής αυτή η ορισμή, σημαίνει πως το πεδίο εφαρμογής ε, των τροπολογιών θα συμπίπτει με την οδηγία περί φορολόγησης ε, τόκων. Και η εισαγωγή στο άρθρο 3α απαιτεί κάποια ερμηνεία, αλλιώς θα έχουμε προβλήματα με την εφαρμογή της οδηγίας. Και συμφωνώ με τους συναδελφούς που είχαν κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά την ε, πρόσβαση σε φορολογικές πληροφορίες. Κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν όλες τις πληροφορίες για όλες τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 8, παράγραφος 1. Πρέπει να τα δούμε και από νομική σκοπιά. Τη συμμόρφωση δηλαδή με συνταγματικές διατάξεις όπως επεσήμανε η street Λούλινγκ όταν είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων υποστήριξα τον εισηγητή μας για να δοθεί μια εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες. Όμως ε, συνειδητοποιώ πως ε, τη λύση αυτή δεν τη στηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη και νομίζω πως ο Ιβο Στρέτσεκ στις τροπολογίες του μας δείχνει μία κατεύθυνση στην οποία θα μπορούσαμε να πάμε. Κάποιοι συνάδελφοι πρότειναν να αναβληθεί η ημερομηνία εφαρμογής. Εγώ είχα κάποιες αμφιβολίες από το Δεκέμβριο του 2014 και παρά το ότι δεν κατέθεσα κάποιες σχετικές τροπολογίες, νομίζω πως πρέπει να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα οι σκιώδεις για να μην βιαζόμαστε. Θα ήθελα να πω πως οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί δεν ε, διαφέρουν τόσο Έχουμε παρόμοιους στόχους ελπίζω να επιτύχουμε συμβασμούς ε, χωρίς ε, άλλη καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κούτας. Ε, λίγα λόγια μόνο να προσθέσω, γιατί δεν ήταν παρόντος οι συνάδελφοι. Είχα πει νομίζω πως είναι καλύτερο να συναντηθούμε στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα για να έχουμε μια σαφή εικόνα για όλες τις τροπολογίες. Και για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σταβάρες συμφωνώ πλήρω Και να δούμε τι συμβαστικές ε, λύσεις ε, θα έχουμε. Για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι στο τέλος. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ. Τελειώνει αυτή η συζήτηση. Να σας πενθυμίσω πως η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας έχει προβληθεί για τις 4 Νοεμβρίου. Εδώ τελειώνουν οι σημερινές εργασίες. Α, κύριος Λάγκεν. Μία παρατήρηση επί της διαδικασίας. Όταν έχουμε Δευτέρες και Πέμπτες ε, συνεδριάσεις τη Επιτροπής μας, σωστό βεβαίω, ε, πρέπει όμως να μην έχουμε ε, Δευτέρα απόγευμα στο Στρασβούργο συνεδριάσεις. Είναι ανεύθυνο την Δευτέρα την επόμενα συνεδριάζουμε μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Έχουμε 8 ψηφοφορίες ε, σε δύο επιτροπές, ΕΚΟΝ και Ήτρε. Και είναι εδώ πέρα οι αίθουσε άδειε τις ε, εβδομάδες ε, των ομάδων. Εγώ δεν έχω έκθεση, ήρθα να δω τι θα γίνει. Αλλά είναι ανευθυνότητα εκ μέρου των συναδέλφων. Δεν γίνεται σωστή κατανομή της εργασίας. Ψηφίζουμε Δευτέρα απόγευμα σημαντικές ε, εκθέσεις και εδώ πέρα έχουμε όσο χρόνο θέλουμε και δεν ασχολείται κανείς. Πρέπει να το δει η Προεδρία. Είτε να καταργηθεί η Δευτέρα απόγευμα του Στρασβούργου, να μην έχουμε ψηφοφορίε τότε, ή ε, αυτή εδώ η αυτη εδω η συνεδριαση Σας ευχαριστώ, κύριε Λάγκεν. Α, τα μεταφέρουμε αυτά θα τα μεταφέρουμε οπωσδήποτε. Επίσης, είμαι 19 χρόνια, 19 χρόνια μέλος αυτής της Επιτροπής. Κάναμε πολλές προσπάθειες να γίνεται σωστά η δουλειά. Αλλά σημαντικά θέματα πάνε Δευτέρα απόγευμα για ψήφιση στο Ρασβούργο, όταν πολλοί συνάδελφοι είναι ακόμη στα μέσα μεταφοράς μέσα. Είναι λάθος. Σας ευχαριστούμε. θα τα μεταφέρουμε στον πρόεδρο της, στην πρόεδρο της Επιτροπής μας. Η ψηφοφορία λοιπόν στις 4 Νοεμβρίου για την έκθεση Κούτας. Η επόμενη συνεδρίαση βλέπετε για, τις, ε, για την Δευτέρα του Στρασβούργου. Ελπίζω να είστε όλοι εκεί. Και μια που είναι η πρώτη φορά εγώ θα χτυπήσω και το σφυράκι. Λίγη τη συνεδρίαση.